με και το Κοινοβούλιο και τα κρατη για τις τελευταίες εξελίξεις. Ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξή σας σε αυτόν τον κοινό μας αγώνα. Ευχαριστούμε. Έχουμε λάβει 7 ε, προτάσεις ψηφίσματος ε, για να κλείσει η συζήτηση και τώρα θα περάσουμε στις ψηφοφορίες. Κυρία Γκόμες, θα σας δώσω το λόγο πριν ε, ψηφίσουμε για την Ινδονησία. Αλλά το επόμενο θέμα είναι η ψηφοφορία για ε, έξι ψηφίσματα σχετικά με την λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Πρώτη τροπολογία με ονομαστική ψηφοφορία η οποία ξεκινά. voted, the vote is now closed. Λίγη ψηφοφορία. Απερίφθη η τροπολογία. Κατόπιν αυτού ε, ψηφίζουμε το ψήφισμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα φαίνεται ότι υπήρξε ένα διοικητικό λάθος σχετικά με τον κανόνα ομιλικτών για την Ινδονησία και γι' αυτό εξαιρετικά θα δώσω τον λόγο στην κυρία Γκόμες για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, έζησα στην Ινδονησία και την αγαπώ. Ξέρω ότι έχει κάνει μεγάλη πρόοδο από τις πρώτες εκλογές το 1999 για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να εκτιμήσουμε και νομίζω ότι αυτό το εκτιμούμε μέσω του ψηφίσματος διότι η Ινδονησία που είναι το μεγαλύτερο μουσουλμανικό κράτος στον κόσμο η μεγαλύτερη ανεξιθρησκεία και σεβασμό των θρησκευτικών πεπιθήσεων. Αν έτσι ενισχύεται η Ινδονησία τότε θα έλεγα μακάρι. Αλλά βλέπουμε ότι και εκεί υπάρχουν ε, ε, διάφοροι ε, διάφοροι ε, ακραίοι, ε, ακραίες δυνάμεις ε, που επιτίθενται κατά τον παππούα, κατά των ιερωμένων και γι' αυτό θα πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση πολιτικά και θα πρέπει να υπάρξει παραδειγματική τιμωρία για να αντιληφθεί η Ινδονησία ότι εμείς ανησυχούμε για τα θύματα και έχουμε πλήρη αλληλεγγύη για όλους τους θαραλέους πολίτες στην Ινδονησία, στην κοινωνία της των πολιτών οι οποίοι μάχονται εναντίον των διακρίσεων και της ατιμορρησίας και θα ήθελα να σας πω ότι η χείρα του ενός ακτιβιστή ε, ο οποίος ε, δολοφονήθηκε προμερικών ετών και όπου δεν έχουν ακόμη δικαστή ε, Ψηφίζουμε υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Τώρα προχωρούμε στην ψηφοφορία για τα έξι ψηφίσματα σχετικά με την Ινδία. και καταρχήν ε, έχουμε ε, το ψήφισμα των ε, Ευρωπαίων Συντηρητικών υπέρ κατά αποχές απερίφθη και τώρα το κοινό ψήφισμα ποιος είναι υπέρ με συγχωρείτε, νομίζω ότι προχώρησα πολύ γρήγορα. Καταρχήν όμως η τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Ε, τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απερίφθη και τώρα το κοινό ε, ψήφισμα ε, με ονομαστική ψηφοφορία η οποία ξεκινά λίγη και εγκρίθηκε. Τα πρακτικά της συνεδριάσεως αυτής θα υποβληθούν στο Κοινοβούλιο προς αποδοχή στην επόμενη συνεδρίαση και ε, κατόπιν αυτού θα προωθήσω τα ψηφίσματα τα οποία ε, υπερψηφίστηκαν και κατόπιν ε,